Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίσω στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας. The following languages are not available today. Danish, Finnish... Δανεζικά, φινικά, φι, φιλαδικά, συγγνώμη, ε, σουηδικά, σλοβενικά και μαλτέζικα δεν είναι διαθέσιμα σήμερα. πρόεδρος της υποεπιτροπής μας δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα και μου ζήτησε να προεδρεύσω αυτή τη συνάντηση που θα, είναι με τη... θα έχει τη μορφή ενό εργαστηρίου. Ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φορέα Άμυνα, θα έπρεπε να έχει έρθει στη συνεδρίασή μας σήμερα στις 9 η ώρα. Λόγω της παρουσίαση του κυρίου Όλι Ρεν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της πρώτης ε, έκθεσης προόδου για τη διεύνηση ακριβώς την ίδια στιγμή έπρεπε εμείς να καταργήσουμε τη συνάντηση με τον κύριο Waze, να την αναβάλουμε για μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Γι' αυτό ξεκινάμε σήμερα στις 10.45. Θα ρέει και στο διαδίκτυο αυτή η συνεδρία. Έχετε παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη. All We continue forward. Εντάξει, συνεχίζουμε προς τα εμπρός. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρούν τα πρακτικά μας ότι έχουν εγκρίθει. Today's workshop on anti-personal landmines η σημερινή μα συνεδρίαση που αφορά τι νάρκες κατά προσωπικού αντανακλά το ενδιαφέρον τη υποεπιτροπή μα για ένα κόσμο χωρί νάρκες κατά προσωπικού. Μετά από τη σύμβαση τη ΟΤΑΒΑΣ που ζητά την πάυση της παραγωγής, ε, αποθήκευση και χρήση ναρκών και φυσικά την καταστροφή των αποθεμάτων που υπάρχουν. Ετέθησε εφαρμογή αυτή η σύμβαση το 1997, έχει επιτύχει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Ορισμένα κράτη όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, Ινδία και Πακιστάν εξακολουθούν να μην έχουν υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Εγώ υπογραμμίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρμαχος αυτής της συνθήκης και ζητά να γίνει οικουμενική και να καλύψει όλα τα κράτη του κόσμου. Αυτό το εργαστήριο είναι πράγματι πολύ επίκαιρο γιατί από τις 30 Νοεμβρίου στις 4 Δεκεμβρίου θα λάβει η χώρα στην Καρταχένα της Κολομβίας μια συνδιάσκεψη για την επισκόπηση της προόδου στο θέμα αυτό. Συνεργαζόμαστε επίσης με τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Δράσεων με στόχο να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε καλύτερα τη δράση όλων των εμπλεκομένων εταίρων σε αυτήν τη διαδικασία. Έχουμε προσκαλέσει λοιπόν τα εξή άτομα. Τον ε, πρεσβευτή Έριξ Βίκρεν, ο οποίος εκπροσωπεί τη Σουηδική Προεδρία, ο κύριος ε, ε, Wigmark από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρεσβευτής κ. Στέφαν Χούση από, την, από το Διεθνές Κέντρο για Ανθρωπιστική Αποναρκοθέτηση της Γενέβης, ο κ. Πίτερ Χέρμπι από την ε, Επιτροπή του Ερθρού Σταυρού και προβελπότησαν δύο επίσης παρεμβαίνοντας ο κ. Φανόρντεν, ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του έργου της Κομισιόν για τα θέματα της αποναρκοθένσης και η κυρία Φραντσίσκα Μπράντνερ, που είναι η εισηγήτρια για το μέσο σταθερότητος, το οποίο είναι σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε πολλά ανθρωπιστικά θέματα και θέματα ασφαλείας. Επίσης υπάρχει και ένα έγγραφο από μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είναι ειδικευμένες στον τομέα της αποναρκοθάτσης, που έχουν εργαστεί σε πολλές περιοχές του κόσμου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν δώσει στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρούμε τώρα με τις παρουσιάσεις που προβλέπονται για αυτό το εργαστήριο. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανοιχτή συζήτηση με παρουσία, με συμμετοχή όλων των μερών, όλων των βουλευτών. Ξεκινούμε με τον κύριο Στέφαν Χιούση, ο οποίος θα παρουσιάσει το, την ομιλία του με τίτλο «Η συνθήκη για την απαγόρευση των ναρκών, κύρια επιτέγματα και τεχνικές πρακτικές για την αντιμετώπιση των ναρκών». Κυρίε και κύριοι, είναι προνόμιο και τιμή για μένα να είμαι μαζί σας σήμερα και να κάνω αυτή την παρουσίαση ενώπιον σας. Λέγομαι Στέφαν Χούζη, είμαι ο Διευθυντής του Κέντρου της Γενέβης για την Ανθρωπιστική Αποναρκοθέτηση. Πρόκειται για ένα διεθνή οργανισμό εμπειρογνωμόνων, ο οποίος έχει την έδρα του στη Γενέβη. Το νομικό της καθεστώς είναι λίγο παρόμοιο με τον οργανισμό του, Εθνικού, του Ερθρού Σταυρού, παρά το γεγονό ότι είμαστε πολύ μικρότερο οργανισμό. Είμαστε ένα ίδρυμα βάσει του ελβετικού δικαίου με διεθνή εντολή. Εμεί έχουμε την ε, γραμματεία κατά κάποιο τρόπο της ε, συνθήκης για την καταστροφή των αρκών με την υποστήριξη των κρατών μελών και της Συντονιστικής Επιτροπής και συγχρόνως έχουμε εντολή να αναπτύξουμε πρότυπα για διεθνεί δράσεις κατά των αρχών που στη συνέχεια θα πρέπει να επικυρωθούν από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και να τύχουν γενικότερη και παγκόσμια εφαρμογή. Ελπίζουμε ότι το κέντρο μα θα μπορέσει να αναπτύξει ένα κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του, της συνθήκης για τα νέα συμβατικά όπλα διασποράς, διότι καλύπτουμε και αυτά τα όπλα και υπάρχει και μια κοινή μεθοδολογία πολλές φορές σε ό,τι αφορά το, το σύνολο όλων αυτών των οπλικών συστημάτων, ιδίως αυτών που δεν έχουν εκραγεί. Θα ήθελα να σταθώ στα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 1999 και εντέφεν, τα τελευταία 10 χρόνια δηλαδή, Μπορώ να πω ότι είναι κάπως ανάμεικτη η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπήρξε σημαντική πρόοδο για την καταστροφή των αποθεμάτων ναρκών κατά προσωπικού. Παράλληλα όμως εξακολουθούν να υπάρχουν πέντε κράτη που έχουν υπογράψει αυτή τη συνθήκη που δεν έχουν ακόμα περατώσει την καταστροφή αυτή. Τρία από αυτά τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, προλάβει την ε, την ε, καταληκτική προθεσμία των τριών ετών η Λευκορωσία, η Ελλάδα και η Τουρκία επίσης του χρόνου δεν θα προλάβει να τελειώσει την καταστροφή των αποθεμάτων. Αυτά λοιπόν για την καταστροφή των αποθεμάτων, αλλά υπάρχουν και όλα τα άλλα κράτη όπως ανέφερα ο πρόεδρος, τα οποία ακόμα δεν έχουν υπογράψει την ε, συνθήκη για την απαγόρευση των αρκών. Σε ό,τι αφορά την αποναρκοθέτηση υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία έχουν αναφέρει ότι έχουν περατώσει τις εργασίες αποναρκοθέτησης, αλλά 19 κράτη που είναι υπογράφοντα τη συνθήκη δεν έχουν ακόμα περατώσει αυτή τη διαδικασία, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μετά από 10 χρόνια εξακολουθούν να έχουν ενεξελίξει ενέργειες ναρκοθέτησης και ζήτησαν παράταση μέχρι και 10 ακόμα χρόνια. 1100 τετραγωνικά χιλιόμετρα ναρκών έχουν αποναρκοθετηθεί και 2.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχών εμπολέμων δράσεων, αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντικέ περιοχέ οι οποίε επηρεάζονται. Αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το γεγονό ότι σε πολλέ από τι χώρε αυτέ υπάρχει επίπεδο ρήπανση το οποίο δεν έχει διακριβωθεί απόλυτα. Ο αριθμό των νέων θυμάτων από τι συνάρκε αυτέ μειώνεται, αλλά όπω γνωρίζετε, από τη στιγμή που υπάρχει ένα θύμα μια τέτοια δράση, ένα θύμα λοιπόν από νάρκες, αυτό το θύμα παραμένει ένα άτομο ανάπηρο που έχει ανάγκες αρρωγής σε όλη του τη ζωή. Πριν από δέκα χρόνια φυσικά ήταν περισσότερα τα ατυχήματα με μη εκραγήσεις νάρκες και ήταν πιο σοβαρό το ανθρωπιστικό πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του προβλήματος που προξενούν αυτές οι νάρκες διότι αποτελούν και εμπόδιο στην ανάπτυξη των ε, αναπτυσσομένων χωρών. Υπάρχουν περιοχές που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία υποδομής, ούτε για γεωργία, επειδή ακριβώς υπάρχουν ενάρκειες στην περιοχή αυτή. να σας αναφέρω μερικά από τα επιτεύγματα και τις μεθόδους που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και που είναι σημαντικές για το μέλλον. Είναι η διαδικασία απελευθέρωσης περιοχών ναρκοθατημένων. Είναι μια συστηματική διαδικασία όπου οι περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες περνάνε μια διαδικασία για να θεωρηθούν ότι είναι απόλυτα ασφαλείς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικονομική ανάπτυξη. Ακολουθούμε μια συστηματική δραστηριότητα, όχι μόνο είχαμε τεχνικές έρευνες, αλλά και μη τεχνικού χαρακτήρα ε, αντιμετώπιση που οδηγεί ένα, ένας χώρος ο οποίος είναι ναρκοθετημένος να καθοριστεί σαφέστερα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά συστήματα για την αποναρκοθέτηση. Σας δίνω ορισμένα στοιχεία για τη Μοζαμβίκη για να καταδείξουν πώς έχει λειτουργήσει αυτή η έννοια της ε, αποναρκοθέτησης και της απελευθέρωσης περιοχών. Μεταξύ του 2000 και του 2002 υπήρξε μια έρευνα για τον αντίκτυπο των αρκών που οδήγησε στο να καθοριστούν 558 τετραγωνικά χιλιόμετρα ως περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες. Μετά από 8 χρόνια <clears throat> από ναρκοθέτησης, μειώθηκαν κατά 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα αυτές τις περιοχές. και βρίσκεται σε επίπεδο μονάχα 500 τετραγωνικών χιλιόμετρων περιοχών που θεωρούνται επικίνδυνες. Στη συνέχεια, μέσα σε ένα χρόνο, με την συστηματική εφαρμογή όλων αυτών των ερευνών και τοπογραφικών αναλύσεων που έγιναν, μπορέσαμε να απελευθερώσουμε σχεδόν 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και να εστιάσουμε την προσοχή μας στα 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα όπου είναι σαφές ότι υπάρχουν επικίνδυνες περιοχές. Ήταν ένα σημαντικό λοιπόν επίτευγμα και είναι και ένα οδηγό για άλλα που θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να γίνει η εκαθάριση των περιοχών αυτών και είχαμε κάποιε επιτυχίε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή η εκαθάριση περιοχών που θεωρούνται επικίνδυνε, βελτίωση στην κατάρτιση, βελτίωση στην πιστοποίηση των σκύλων που χρησιμοποιούνται στην αποναρκοθέτηση, καλύτερη δοκιμασία των μηχανισμών αποναρκοθέτησης και ένα σύνολο από τεχνικό εξοπλισμό που υπάρχει στην αγορά για να αντιμετωπίσει τις ενέργειες αποναρκοθέτησης. Θεωρώ όμως ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει σημαντική πρόοδος με καλύτερη διαχείριση των προγραμμάτων και όχι περισσότερο μέσω τεχνικής βελτίωσης. Έχουμε φτάσει ήδη σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ικανότητας. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον Τεκ Πάτερσον, ο οποίος είναι ο επικεφαλής οικονομολόγος στο κέντρο μας, ο οποίος έχει κάνει και την αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποναρκοθέτηση. Σας, Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να θίξω αυτά που ανέφερε ο πρέσβης Χούζη για τις σταθερές ε, που εφαρμόζει τι τεχνολογικές καινοτομίες αλλά και ακόμη πιο σημαντικό στη διαχείριση των καινοτομιών σε αυτόν τον κόσμο που συχνά αποκαλείται ανθρωπιστικό όσον αφορά την ε, εξουδετέρωση των ναρκών. Έχουμε να κάνουμε με δύο εκαθαρίσεις, δύο ειδών εκαθαρίσεις από στρατιωτικές μονάδες ή από ομάδες πολιτών ε, στην ίδια χώρα κατά τη διάρκεια της ίδιας ειρηνευτικής διαδικασίας. Και δείχνουμε, βλέπουμε ότι η αποναρκοθέτηση από τις ομάδες των πολιτών είναι 60 με 65 φορές λιγότερο δαπανηρό από ότι η αποναρκοθέτηση από τους ε, στρατιωτικούς. Ως αποτέλεσμα, οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ όλες εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ για τις ε, δράσεις κατά των ναρκών, ώστε να μπορούν να καλούν πολίτες για την επαναρκοθέτηση, για την υποστήριξη των στόχων των ε, αποστολών μας, που είναι όλες ειρηνευτικές. Έχουμε επίσης το προνόμιο να διεξάγουμε μελέτες, ε, τα έξι περιφερειακές μελέτες, για τις ε, δράσεις επανορκοθέτησης ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτούνται από το 2002 μέχρι το 2007. Πλαίσιο των μελετών αυτών ήταν ότι υπήρχαν δύο στρατηγικές ε, για δράσεις για τις νάρκες που ζητήθηκαν από τους κανονισμούς που υιοθέτησε το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Και για τις νάρκες κατά προσωπικού και για τους μη για τους εξοπλισμούς που δεν έχουν εκραγεί. Οι στρατηγικές αυτές υποστηρίχθηκαν από την γραμμή του προϋπολογισμού με, για την ε, σνάρκης κατά προσωπικού με 15 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο, πρώτο τρίμηνο και 60 για το υπόλοιπο του χρόνου. Για να σας συνοποιήσω σύντομα, η στρατηγική ήταν ε, πολύ επιτυχής και οι στόχοι επετεύχθησαν. Οι μεταρρυθμίσεις ε, στο σύστημα ε, ενισχύσεων του 2006 οδήγησαν στην εξάλληψη του θεματικής γραμμής για την εξουδετέρωση των αρκών κατά προσωπικού. Ε, στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Έπειτα, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις για τις νάρκες που κατευθύνουν τις αντιπροσωπείες ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες που ήταν τώρα πιο υπεύθυνε για το προγραμματισμό και τον καθορισμό των προγραμμάτων αλλά και την υποπτία αυτών είναι ένα μεγάλο έγγραφο το οποίο όμως δεν αντισταθμίζει τη συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού καθώς και τα συμπληρώματα ε, από τις νάρκες κατά προσωπικού. Σε αυτή τη φάση, αυτή τη χρονική στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προγραμματισμός καθώς και το σύστημα αποτελεσμάτων σε σχέση με τις δράσεις ε, του, για τις νάρκες είναι πολύ αποκεντρωμένος. Υπάρχουν γεωγραφικές γραμμές του προπολογισμού που έχουν στόχο την αποναρκοθέτηση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στις πολύ ε, ναρκοθετημένες χώρες θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένους φαγγέλους, όπως το Αφγανιστάν για παράδειγμα ή η Αγγόλα, διότι διαφορετικά δεν γίνεται να ανταποκριθούμε στις ανάγκες άλλων χωρών σε σχέση με την αρποναρκοθέτηση. Ε, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που χρηματοδοτούνται λιγότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Καμπότζη. Δεν υπάρχει μηχανισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει διεθνείς δράσεις. Γίνονται όλα ανά χώρα και η απώλεια της θεματικής γραμμής του προπολογισμού οδήγησε, ε, συνοδεύτηκε μάλλον και με, από μία μείωση του προσωπικού ε, και άρα απώλεια εμπειρογνωμοσύνης στα αρμόδια όργανα και άρα και κανένας μηχανισμός για να προϋποστηριχτούν παγκόσμιες ή περιφερειακές πρωτοβουλίες με στρατηγικό τρόπο. Έχουμε λοιπόν διάφορες συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προγραμματισμό και την δράση για τις νάρκες. Εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή προϋπολογισμού ή συγκεκριμένους... Ε, μηχανισμός για τη χρηματοδότηση των δράσεων κατά των ε, ναρκών αλλά και των ε, των βομβών διασποράς ε, μπορεί να πετύχουμε κάποια πράγματα αλλά λιγοστά με περισσότερες δαπάνες και με πιο συνεκτική προσέγγιση θα χρειαζόταν μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη από τις Βρυξέλλες, που υπάρχει στις Βρυξέλλες, για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε με παγκόσμιο και στρατηγικό, στρατηγική μάλλον προοπτική. Σας ευχαριστώ. The floor for Mr. Peter Herby. Το λόγο έχει ο κύριος Πίτερ ε, στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού. Στη Γενέβη φυσικά. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να έρθω ενώπιόν σας και εσάς και άλλους συναδέλφων και ε, με ενδιαφέροντες ε, οργανισμούς. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερθρού Σταυρού ασχολείται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας 90 με αυτά τα θέματα των αρκών κατά προσωπικού. Όταν διαπιστώσαμε ότι από μόνο του αυτό το όπλο ε, δημιούργησε επιδημία ε, τραυματισμών από νάρκες, όπως το χαρακτηρίζει το ιατρικό μας προσωπικό, παντού στον κόσμο, σε εμπόλεμες ζώνες. Πώς σταματάει η επιθυμία. Για να σταματήσει μια επιθυμία θα πρέπει να ε, καταπολεμηθεί στη ρίζα της, στην αιτία του κακού. Αυτά οι ε, νάρκες είναι μικρά οπλικά συστήματα, υπάρχουν παντού και κάνουν τεράστιες ζημιές παντού όπου ε, χρησιμοποιούνται κυρίως σε άμαχο πληθυσμό μετά τον πόλεμο και όχι σε στρατιώτες κατά τη διάρκεια της σύραξης. Αυτά ε, είναι η, τα θεμέλια, τα ανθρώπινα και τα ανθρωπιστικά. Η Σύμβαση της Γενέβης είναι από τις τη συνθήκη μάλλον για την απαγόρευση ε, είναι ε, από τις πιο επιτυχημένες διεθνώς για πολλούς λόγους. Δέκα χρόνια και πλέον μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης διαπιστώνουμε ότι παραμένει πάρα πολύ επίκαιρη, πάρα πολύ δυναμική και πάρα πολύ επίκαιρη και ε, προοδεύει και εφαρμόζεται. Δεν είναι μόνο στα χαρτιά μια σύμβαση, αλλά ένα πρόγραμμα για να πετύχουμε επιτόπου ένα ανθρωπιστικό στόχο. Εγώ θα εξτάσω τα θέματα κυρίως ε, με βάση της διάσκεψης αναθεώρησης της Καρθαγένης που θα γίνει σε έξι εβδομάδες. Η δεύτερη, η πρώτη ήταν στο Ναϊρόμπι το 2004 και κατήρτισε και το πρόγραμμα δράσης του Ναϊρόμπι. Στην Καρθαγένη θα έχουμε το πρόγραμμα της Καρθαγένης που θα ορίσει το επόμενο πενταετές ε, πλαίσιο. Να σας αναφέρω πρώτα τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα. Ο πρέσβης ε, κύριος Ιουσί ε, ανέφερε και μερικά και σύντομα στη συνέχεια θα σας αναλύσω τις ε, προκλήσεις του μέλλοντος που είναι πλέον πολύ σαφέστερες από τη... στην πρώτη αναθεώρηση το 2004. Ας αρχίσουμε από τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πιστεύω, ότι 156 χώρες είναι συμβαλόμενα μέρη, πάνω από τα 3 τέταρτα του συνολικού ε, αριθμού κρατών. Επίσης έχει στιγματιστεί η χρήση ε, ναρκών κατά προσωπικού από τον καθένα και παντού. Αυτό ξέρετε έχει και αντίκτυπο ε, στην τακτική και στην πρακτική των μεγάλων δυνάμεων που παραμένουν εκτός. Μεταξύ αυτών και οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1991 δεν χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα και η Ρωσία και ε, η Κίνα που έχουν απαγόρευση εξαγωγών εδώ και 10 και πλέον έτη. Και χώρες ακόμα όπως το Πακιστάν που έχουν ε, μαζικά ναρκοθετήσει τα σύνορά τους προς το Αφγανιστάν ε, τελικά επηρεάζονται και από τα διεθνή τεκτενόμενα για να μην προχωρούν σε αυτή την ναρκοθέτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αποναρκοθέτηση, ε, ε, χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ναρκοπεδίων έχουν καθαριστεί με επίπονο τρόπο εδώ και χρόνια και αλευθερώθηκε γη για παραγωγική δραστηριότητα και βεβαίως ε, προελήφθηκαν και νέα θύματα από νάρκες. Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση και καταστροφή τους, μέχρι το 2008 ε, είχαν από ε, αποθέματα ε, τα κράτη και τρία από αυτά δεν τα κατέστρεψαν. Θα έρθω σε συνέχεια σε αυτό. Γενικά καταστράφηκαν 42 εκατομμύρια νάρκες κατά προσωπικού που ποτέ δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση. Ε, η σύμβαση πώς ξεκίνησε. Από την ανησυχία για τα δεινά που υποφέρουν τα θύματα ε, ε, και επικεντρώθηκε στο πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές. Τελικά είχαμε κινητοποίηση ορισμένων αλλά όχι αρκετών ε, πόρων για παροχή βοήθειας στα θύματα. Τώρα, ε, σε σχέση με την προστασία και τη βοήθεια των θυμάτων δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα θύματα από τις νάρκες κατά προσωπικού, αλλά θα τους βοηθήσει στο δινικές αυτό αργότερα. Αυτή λοιπόν η παροχή βοήθειας στα θύματα έχει κατοχυρωθεί ε, και σε ολόκληρη παράγραφο για αντίστοιχη σύμβαση που διέπει τα ε, όπλα αυτά. Έχει γίνει λοιπόν κανονικό άρθρο με ε, νομικά δεσμευτική ισχύ στις βόμβες διασποράς και την αντίστοιχη σύμβαση για αυτές. I think it's, it's also quite significant. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά την θέση σε εφαρμογή αυτής της σύμβασης υπάρχουν επαφές μεταξύ των συμβαλωμένων μερών για να, δούμε, για να δουν πώς γίνεται η εφαρμογή της σύμβασης αυτής δύο φορές κάθε χρόνο τα τελευταία δέκα χρόνια και προβλέπουν να συνεχίσουν αυτές οι επαφές τα επόμενα πέντε χρόνια. Αν δείτε άλλες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό των όπλων τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει κάποιο άλλο καθεστώς το οποίο είναι τόσο δυναμικό και το οποίο έρχεται συνέχεια σε αντιπαράθεση με τις υποχρεώσεις του όπως αυτό για την απαγόρευση των ναρκών. Τα περισσότερα άλλα συστήματα έχουν το πολύ μία ετήσια συνάντηση μεταξύ των συμβαλεμένων μερών και το πολύ πέντε συνδιασκέψεις αναθεώρησης. Υπάρχει λοιπόν μια ποιοτική διαφορά μεταξύ της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Αρκών, η οποία είναι πραγματικά στρατευμένη στην ε, αντιμετώπιση των αρκών έναντι άλλων συμβάσεων που υπάρχουν με απαγορεύσεις αλλά δεν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της πρόοδου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά αυτήν την ε, σύμβαση, αντίθετα με άλλες ανθρωπιστικές συνθήκες και συμβάσεις, δεν είναι μονάχα μια απαγόρευση χρήσης ναρκών, αλλά και μια σύνολη διαδικασία, ένα πρόγραμμα δράσης για την αποναρκοθέτηση και την καταστροφή των ναρκών για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο ανθρωπιστικό αποτέλεσμα. Αν στραφώ τώρα στις προκλήσεις ενώπιών μας. Μετά από δέκα χρόνια εφαρμογής της σύμβασης είναι σαφείς οι προκλήσεις Νομίζω ότι η συνδιάσκεψη της Καρθαγένης θα παίξει ένα κομβικό ρόλο για να καθορίσει το κατά πόσο αυτές οι προκλήσεις θα τύχουν αντιμετώπισης, αν θα δημιουργηθεί μια κουλτούρα συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη συνθήκη, αν θα διατηρηθεί αυτή η κουλτούρα και αν πράγματι η σύμβαση αυτή θα επιτύχει πλήρως τους στόχους που έχει θέσει στον εαυτό της. Σε ό,τι αφορά την αποναρκοθέτηση. Από τις 21 χώρες οι οποίες είχαν προθεσμίες από ναρκοθέτης που εξέπνεαν πέρσι ή μάλλον φέτος, 15 ζήτησαν παράταση από 1 έως 10 χρόνια, οι περισσότερες αιτήσει ήταν για παράταση δεκαετή. Κατά την άποψή μας αυτό είναι ατυχές. Η σύμβαση επέτρεπε να υπάρχει μια παράταση για τη βασική καταληκτική προθεσμία των 10 ετών, αλλά η δέσμευση που ανέλαβαν όλα τα κράτη-μέλη ήταν να προχωρήσουν στην αποναρκοθέτηση το ταχύτερο δυνατό. Πολλά από τα κράτη που είχαν αναλάβει τη δέσμευση αυτή ξεκίνησαν συγκεκριμένε δράσει ή ακόμα και την αντιμετώπιση της ε, έκταση του προβλήματο μόνο ένα ή δύο χρόνια πριν από μόνο ένα ή δύο χρόνια πριν από την καταληκτική προθεσμία. Γι' αυτό τόσα πολλά συμβαλόμενα μέρη ζήτησαν παράταση τη παρα... της προθεσμίας. Χώρες η Καμπότζη, η Αγκόλα, το Αφγανιστάν θα χρειαζόταν πάνω από 10 χρόνια. Αυτό ήταν εύλογο. Και θα χρειαζόταν και την βοήθεια άλλων κρατών και θα ήταν ένα τρόπο αυτό να δώσουν περισσότερη έμφαση στα προβλήματά τους και να κινητοποιήσουν πόρους και από απ' έξω για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Αλλά αυτό δεν προβλεπόταν για χώρες οι οποίες απλώς είχαν ναρκοπαίδια στρατιωτικού χαρακτήρα και μερικές δεκάδες χιλιάδες ναρκών και μετά από 10 χρόνια εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα αυτά τα ναρκοπαίδια. Όχι λοιπόν για χώρες με μικρά προβλήματα που μόνο την τελευταία στιγμή, 8 χρόνια μετά την υπογραφή της συμβάσεως, άρχισαν να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι μια τάση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και την αναστρέψουμε. Εάν δεν την αντιμετωπίσουμε, μερικές από τις χώρες που έχουν τύχη παράτασης θα ζητήσουν και περαιτέρω παρατάσεις, κάτι το οποίο θα υποσκάψει την πορεία της σύμβασης αυτής, δεν θα είναι καλό μήνυμα και θα σημαίνει ότι ο αντίκτυπος αυτών των ναρκών και τα ανθρώπινα βάσανα που προκαλούν θα εξακολουθούν να υφίστανται. Σε ό,τι αφορά την καταστροφή των οπλοστασίων και εκεί δυστυχώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου τρεις χώρες δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν την καταληκτική προθεσμία που δεν επιδέχεται παράταση και επομένως έχουν παραβιάσει τις ε, προθεσμίες. Είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Λευκορωσία και η Ουκρανία επίσης έχει ανακοινώσει ότι δεν προβλέπει να μπορέσει να προλάβει αυτή την προθεσμία που εκπνέει το Μάρτιο του 2010. Τέσσερις χώρες στην περίπτωση της Ελλάδος και της Τουρκίας με αποθέματα ενός εκατομμυρίων ναρκών κατά προσωπικού, 3 εκατομμύρια για την ε, Μπελαρούς, 6 εκατομμύρια για την Ουκρανία. Δεν έχουν καλύψει λοιπόν την προθεσμία τους, αυτό είναι πραγματικά μια περίπτωση μη συμμόρφωσης με το κείμενο της σύμβασης. Μπορεί να υπάρχουν <clears throat> πολλοί λόγοι για του οποίου οι χώρε αυτέ δεν έχουν συμμορφωθεί με την προθεσμία. Μεταξύ των άλλων, στην περίπτωση τη Μπελαρού, τη Λευκορωσία δηλαδή και τη Ουκρανία, υπάρχουν λόγοι που οφείλονται στο πολύπλοκο έργο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία δεσμών χρηματοδότησης για τα θέματα αυτά όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέτρινε την ε, Λευκορωσία και την Ουκρανία να κυρώσουν τη σύμβαση αυτή και το έκαναν αυτό με τη ρητή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα δώσει χρηματοδότηση για την καταστροφή του οπλοστασίου ναρκών και πιστεύω ότι θα ακούσετε περισσότερα από την Κομισιόν για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, χρειάστηκε διαπραγματεύσεις, διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών που εγώ δεν μπορώ να πω ότι τις κατανοώ, αλλά σίγουρα ήταν αργές και πολύ πιο επίπονες από ό,τι περιμέναμε. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τέσσερα κράτη με περίπου 12 εκατομμύρια ενάρκειες κατά προσωπικού που αποτελούν μια παραβίαση των ε, προθεσμιών που είχαν τεθεί. Αυτό είναι μια παραβίαση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εμείς ενθαρρυνόμαστε από αυτά που ακούσαμε για την πρόοδο που έχει γίνει τόσο από τη Λευκορωσία όσο και από την Ουκρανία για τις διαπραγματεύσεις που έχουν κάνει με την Κομισιόν. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι οι χώρες αυτές θα μπορέσουν στην ε, διάσκεψη αναθεώρησης της Καρθαγένης το πώς και πότε θα μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους για την καταστροφή των μεγάλων προστασίων που έχουν και τελικά αυτά είναι θέματα που έχουν μείνει στο εδαφός τους μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν είναι καν λοιπόν οπλοστάσια λευκορωσικά ή ουκρανικά. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την αρρωγή προς τα θύματα. Παρά την ε, γενικότερη κατανόηση που επετεύχθη και την καλύτερη εστίαση επί του πρακτέου, η επιτόπια πραγματικότητα στις περισσότερες χώρες και για τα περισσότερα θύματα ναρκώνουν ότι λίγα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Η Handicap International, μια οργάνωση που ασχολείται με τα θέματα αυτά είχε δημοσιεύσει πρόσφατα μια έκθεση που βασιζόταν σε συνεντεύξεις με 3.000 περίπου θύματα από όλο τον κόσμο και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα θύματα αυτά και οι κοινότητες τις οποίες ζουν δεν έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης, ιατρικές υπηρεσίες αποκατάστασης τα τελευταία 10 χρόνια. Σε ορισμένε περιπτώσεις η εμπειρία ήταν ότι η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος των δεκαετών και αυτό φαίνεται και από την εμπειρία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Υπήρξαν περιοχές όπου τα πράγματα βελτιωθήκαν, υπήρξαν ευρύτερα προγράμματα ορθοπαιδικής αποκατάστασης που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά εισάριθμος αριθμός περιοχών και χωρών όπου τα προγράμματα αυτά έχουν πάψει να λειτουργούν λόγω έλλειψης πόρων ή θέλησης. Θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχει μια έκκληση που έχει δοθεί σε όλα τα κράτη τα οποία συμμετέχουν στην συνάντηση της Καρθαχένης. Αυτό είναι <clears throat> τα πορίσματα των ατόμων που πρακτικά επί το οποίο προσπαθούν να βοηθήσουν τα άτομα τα έχουν τραυματιστεί από νάρκες και οι οποίοι συναντηθήκαν τον Ιούνιο στο Όσλο και ένα από τα πιο στεναρά στοιχεία αυτής της έκκλησης, όπως αναφέρεται και από τους ίδιους, είναι ότι οι περισσότεροι επιβιώσαντες από ατυχήματα μενάρκες δεν έχουν τύχει ακόμα βελτίωσης στην περίθαλψή τους και στην προσωπική τους ζωή. Είναι δύσκολο να καταμετρήσουμε ακόμα την πρόοδο για τα θέματα αυτά. Η διάσκεψη της Καρθαγένης για ένα κόσμο χωρίς νάρκες θα πρέπει να είναι ένα σημείο καμπής, ένα σημείο που αρχίζει να αλλάζει αυτή η πραγματικότητα και αυτή η συνάντηση του Όσλο επίση έχει δώσει συστάσει για το πώ πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Σίγουρα όμω πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αρρωγή προ τα θύματα των αρκών. Αυτό μα φέρνει τέλο στο θέμα των πόρων που ουσιαστικά διατρέχει όλες αυτές τις προκλήσεις που ανέφερα. Την, ε, οι καταληκτικές προθεσμίες βασιζόντουσαν στο στην υπόθεση ότι θα υπήρχε διπλασιασμός, τριπλασιασμός ή και πενταπλασιασμός των απαραίτητων πόρων για να καλυφθούν οι καταληκτικές προθεσμίες. Χωρίς αυτούς τους πόρους δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Η καταστροφή του οπλοστασίου, τουλάχιστον στην περίπτωση της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, είχε προβλήματα πόρων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι στο μέλλον θα υπάρξει κάποια συγκεκριμένη βελτίωση μετά από την καθαγέννη. Η αρρωγή προς τα θύματα εξακολουθεί να είναι θέμα το οποίο εξαρτάται από τους πόρους. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει μονάχα με τα θύματα των ε, <clears throat> ναρκών, αλλά και δημιουργίας υποδομής ιατρικής περιοχής περιοχές που υπάρχουν τα περισσότερα ατυχήματα προς ε, όφελος των θυμάτων και των οικογενειών τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο σχετικά. Και κάτι ακόμα το οποίο έχει προτείνει ο Διεθνής η Ερυθρός Σταυρός και η Ζάμπια είναι να δημιουργηθεί ένας μόνιμος φορέας ο οποίος θα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα των θυμάτων στο μέλλον με πιο συστηματικό τρόπο δηλαδή να τα αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό θα ήταν μια ευκαιρία και για, τους, για τα συμβαλόμενα κράτη που δεν είχαν κατανοήσει το πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν είχαν ένα τέτοιο μόνο φορέα θα είχαν μεγαλύτερε δυνατότητε να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταβατικό αυτό διάστημα. Επίση, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη ε, καταστροφή των αρκών ω θέμα ανάπτυξη. Επομένω, να συμπεριλάβουμε όλε τι οπτικέ γωνίε και όλε τι πτυχέ του θέματο αυτού μια σειρά ενεργειών για την κινητοποίηση των πόρων τα πρώτα πέντε χρόνια. Στη συνέχεια πέρασε η έμφαση στην χρήση των πόρων. Αυτό όμως έχει και μια απόχρωση συγκεκριμένη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινά όλες αυτές οι πτυχές του θέματος. Εν κατακλείδη λοιπόν η συνδιάσκεψη αναθεώσεις καθαχένης θα παίξει κομικό ρόλο για το πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα και πώς θα συνεχιστεί η εφαρμογή της ε, σύμβασης της ΟΤΑΒΑς. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα και τα ζητήματα μη συμμόρφωσης και τα ζητήματα περαιτέρω από ναρκοθέτησης και εκαθάρισης τονίζοντας τη νομική υποχρέωση να γίνει αυτή η εκαθάριση το ταχύτερο δυνατό και όχι μόνο όταν προσεγγίζουν οι καταληκτικές προθεσμίες που οδηγεί πολλού να το κάνουν αυτό μοναχά την τελευταία στιγμή. Επίσης χρειάζεται μια δέσμευση για καλύτερη αρρωγή προς τα θύματα. Και εν κατακλείδη θέλω να τονίσω ότι οι, τα πρότυπα που έχουν τεθεί από αυτή τη σύμβαση είχαν ευρύτερες επιπτώσεις παρά μόνο την αντιμετώπιση των ναρκών κατά προσωπικού. Επίσης, απετέλεσε και πρότυπο για την αντιμετώπιση των οπλισμών διασποράς κατά του άμαχου πληθυσμού και αυτό οδήγησε στην υπογραφή μιας σύμβασης από 100 χώρες που μάλλον θα τεθεί ε, σε εφαρμογή του χρόνου για τα όπλα διασποράς και αυτό θέτει νέα πρότυπα για ένα όπλο το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και ανθρώπινα βάσανα σε όλες σχεδόν τις περιοχές όπου χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα. <clears throat> Επίσης, το ίδιο συμβαίνει για τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της, ε, των σειράξεων και μετά από τις ε, σειράξεις για τα μη εκραγέντα συμβατικά όπλα. Και υπάρχει το πρωτόκολλο για τα όπλα αυτά που προβλέπει δεσμεύσει των κρατών που συμβάλλονται για την πρόληψη της έκρηξης αυτών των όπλων και την μεταγενέστερη εκαθάρισή τους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει τώρα ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, ένα ήπιο αν θέλετε πρότυπο σε διεθνές επίπεδο που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση όπλων που εξακολουθούν να είναι θανατηφόρα όπως τα λέμε. Δηλαδή όπλων που μετά από τη χρήση τους επί δεκαετίες μπορούν να σκοτώνουν ανθρώπους ακόμα και αν δεν εξυπηρετούν κανένα στρατιωτικό στόχο. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν δεσμεύσει στον τομέα της πρόληψης, απαγόρευση των όπλων αυτών όταν δεν φτάνει η πρόληψη και αυτό αφορά τις νάρκες και τα όπλα διασποράς και επίσης την αρρωγή των θυμάτων. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια ιστορική εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε για τα αποτελέσματα των εκρηκτικών οπλισμών που χρησιμοποιούνται σε σειράξεις. Μετά από την ε, εφεύρεση του δυναμίτη, τα όπλα τα οποία τα μη εκραγέντα όπλα που παρέμεναν μετά από μια ένοπλη σύραξη ήταν ουσιαστικά θέμα των τοπικών κοινοτήτων όπου βρισκόντουσαν αυτά τα όπλα. Και αυτό σήμαινε μεγάλους κινδύνους για αυτές τις τοπικές κοινότητες. Τώρα είναι κάτι το οποίο απασχολεί τη διεθνή κοινότητα και θεωρούμε όλοι ότι δεν είναι επαρκές να αφήνουμε την τοπική κοινότητα να τα βγάλει πέρα και βασίζεται στην ιδέα ότι οι χρήστες αυτών των όπλων έχουν μια πολιτική και ηθική υποχρέωση να προλάβουν τα θανατηφόρα αποτελέσματα αυτών των αρκών και να αντιμετωπίσουν τα θύματά τους με έναν τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τα ανθρώπινα βάσανα από τη χρήση αυτών των όπλων. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χέρμπι, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Βίγνερ, συντονιστής ε, για τις Νάρκες στο Σουηδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας για την πρόσκληση που απευθύνατε στη Σουηδική Προεδρία για τη σημερινή ακρόαση. Και για την Προεδρία όπως και για άλλους, τώρα η σημασία ε, και η προσοχή εστιάζεται στη δεύτερη αναθεώρηση της Καρθαγένης και συνεργαζόμαστε με τον Ορβηγό Πρόεδρο, πρέσβη Έκε και συζητούμε τις διάφορες δηλώσεις και τα διάφορα έγγραφα που θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη διάσκεψη αυτή καθώς θα αποτελέσουν το τελικό έγγραφο. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλώ για τη δεύτερη ε, προπαρασκευαστική επιτροπή, που συνεδρίασε αρχές Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε μόνο μερικά γενικά σχόλια. Σε αυτά θα επιμείνω και στη συνέχεια θα σας αναφέρω και κάποιες άλλες σκέψεις. Στη δήλωσή μας Υποστηρίζουμε πλήρως τις προετοιμασίες ε, του πρέσβη Χέκ, όπως και άλλοι διαπιστώνουμε και εμείς ε, ότι έχει γίνει πρόοδος ε, για να δοθεί παγκόσμια διάσταση στη συνθήκη και να ενισχυθεί και ίδια. Επιμένουμε στις προκλήσεις όμως και τις ε, ανθρωπιστικές και ε, τις ε, υπόλοιπες που απορρέουν από τις νάρκες που βρίσκονται σε ναρκοπαίδια. Είναι βασική προτεραιότητα λοιπόν η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα. Επίσης είπαμε ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία δεκαετία στη σύμβαση δείχνει πόσο μεγάλη είναι η στράτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δίνουν περίπου τη μισή χρηματοδότηση παγκοσμίω όλη αυτή την περίοδο για την καταπολέμηση των αρκών. Καλωσορίζουμε λοιπόν ε, το γενικό κορμό των προτάσεων ε, των εγγράφων ε, του Νορβηγού Προέδρου και πραγματικά το θέτουμε το κέντρο βάρου στο ανθρωπιστικό τομέα. Θα πρέπει να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη και να βελτιώνονται οι ζωές ε, των θυμάτων και των κοινοτήτων στις οποίες ζουν. Τα θύματα των αρκών κατά προσωπικού θα πρέπει να συμμετέχουν επίσης, να ακούγεται η φωνή τους. Αυτό το δίδαγμα ε, φάνηκε από μία μελέτη. Μία διεθνή μελέτη που ανέβαινε και ο Πίτερ Χέρμπι προηγουμένως. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων στην κοινή δράση που αποφασίστηκε πέρυσι το 2008, προχωρεί σε ε, κάποιες ενέργειες. Είναι μια κοινή δράση που θα ισχύσει μέχρι την επόμενη άνοιξη και μιλά για ε, περιφερειακά σεμινάρια, τεχνικές επισκέψεις, ε, επιτρέπει σε ε, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, πολύ σημαντικό αυτό, να συμμετέχουν και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και διδάγματα έτσι ώστε να ε, προάγεται η ε, εφαρμογή και η συμμόρφωση αλλά και η παγκόσμια διάσταση του θέματος αυτού. Από την κοινή αυτή δράση έχουμε διαμορφώσει κάποια γνώμη και ε, εντύπωση και θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη καλά θα κάνουν να σκεφτούν πώς θα δώσουν συνέχεια στην κοινή αυτή δράση όταν ε, εκπνεύσει του χρόνου η ισχύουσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης τονίζει συνεχώς τις προσπάθειες που γίνονται για να επικρατήσει παγκοσμίω η σύμβαση αυτή. Είπαμε ότι τα συμβαλώμενα μέρη σήμερα είναι 156, αλλά λείπουν πολλές ε, σημαντικές χώρες. με τους κανόνες και τις προδιαγραφές συμφωνούν όλοι. Και είναι σπάνια η χρήση των αρκών κατά προσωπικού σήμερα. Από την άλλη όμως ε, υπάρχουν οπλοστάσια, υπάρχουν αποθέματα και κάποιοι μη κρατικοί φορείς ε, ε, τις χρησιμοποιούν και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Όπως ακούσαμε έχει γίνει πρόοδο στην αποναρκοθέτηση και στην καταστροφή των αποθεμάτων, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν. Ορισμένες χώρες ε, ήδη παραβιάζουν το άρθρο 4 για την καταστροφή των αποθεμάτων και αυξάνεται ο αριθμός των κρατών εκείνων που ζητούν ε, παρατάσεις Όπως ακούσαμε, 70 χώρες έχουν ακόμα ναρκοπαίδιο στο έδαφος Και η περισσότερη γνώση που έχουμε είναι από ε, την οργάνωση, τον οργανισμό ICBL που καλύπτει διεθνώς αυτά τα θέματα και υπάρχει και ένα παρατηρητήριο ε, για τις νάρκες ε, που δημοσιεύει μελέτες και συμμετέχουν και υποστηρίζουν και η Σουηδία και πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το σχέδιο προγράμματος δράσης που συζητούμε αυτό το διάστημα, όπως ακούστηκε προηγουμένως, Είναι σημαντικό οι προσπάθειε ε, παροχή ε, βοήθειας στα θύματα να εντάσσονται σε ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται εκεί και σχέδια δράσης για αντιμετώπιση παγκοσμίω. Ένα άλλο θέμα που τόνισε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δήλωσή της είναι κάτι σχετικό με αυτό που είπε ο Πίτερ προηγουμένως για τα άλλα ε, νομικά μέσα που θα πρέπει να διερευνήσουμε αν ε, υπάρχει δυνατότητα συνέργειας μεταξύ αυτής της σύμβασης και άλλων ε, συμβάσεων όπως εκείνη για τις βόμβες διασποράς ή τα πυρομαχικά διασποράς και το άρθρο 5 της σύμβασης για τα συμβατικά όπλα. Ολοκληρώνοντα λοιπόν και συμπερασματικά θα πρέπει να σας πω ότι η Προεδρία προσβλέπει στην αναθεώρηση της Καρθαγένης και στη διάσκεψη αυτή ως ευκαιρία να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των ενεχομένων κρατών και να υπάρχει καλύτερο συντονισμός ε, των δωρητών, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ε, καταστροφή και στην αποναρκοθέτηση και όλα αυτά τα θέματα που ανέφερε προηγουμένως ο πρέσβης κύριος ε, ε, Χούση για τη βελτίωση ε, των μεθόδων και της διαχείρισης. Οι νάρκες κατά προσωπικού, τα υπολείμματα βομβών διασποράς οφείλουν, ευθύνονται για πολλά θύματα, έχουν πολλές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες και δεν ε, επιτρέπουν σταθεροποίηση, συμφιλίωση και οικονομική επανάκαμψη. Και επίσης πλήττει τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσει να εστιάζει την προσοχή της εκεί και να συμπεριλαμβάνεται στην αναπτυξιακή της πολιτική πάντα και η δράση αυτή ε, της αποναρκοθέτησης και της καταπολέμησης των αρκών τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δράση της κατά των ναρκών για την επόμενη πενταετία τονίζονται όλα αυτά τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε κατά τα άλλα ε, τον προηγούμενο μήνα ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο προετοιμάζοντας ε, ε, τη διάσκεψη αυτή και συζήτησε όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί στην Καρθαγένη για το ε, πώς δηλαδή θα βελτιωθεί η κοινή δράση και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thanks. And now... Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Βίτμαρ που είναι επικεφαλής ε, του Τμήματος ε, Πολιτικής Ασφάλειας της ΡΕΛΕΞ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να σας κάνω πολύ σύντομα μια παρουσίαση. Ορισμένα από αυτά τα σημεία ήδη αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους από τη Γενέβη, οπότε ταυτόχρονα θα προσπαθήσω να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις ε, από αυτές που εθίγησαν. Η συνάδελφος Μαρία Κρούστη Κριστομπάλ, άμα βρει το σωστό σημείο για να κάνει κλικ, θα μας δείξει και τις διαφάνειες και είναι μάλιστα ο άνθρωπος ε, για την επαφή στη Ρελέξ για όλα τα θέματα ναρκών. Και αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, στραφείτε σε εκείνην. Ενώ αναζητώνται οι σωστές διαφάνειες, να σας πω πως έχουμε ένα σύστημα τώρα στην Κομισιόν ώστε να διασφαλίσουμε πως οι κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες αναφέραμε ε, ακολουθούνται. Έχουμε λοιπόν σημεία επαφής σε ολόκληρη την οικογένεια ρελέξ, διότι οι δράσεις για τις νάρκες είναι κάτι, όπως ήδη υπόθηκε, που αποτελεί τμήμα διαφόρων γεωγραφικών και περιφερειακών προγραμμάτων. δύο το δύο διαφάνεια δύο παρακαλώ. Έχουμε τέσσερα τμήματα σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Να σας δώσω το γενικό πλαίσιο, Κάποια αρχέ κλειδιά και κάποιους μηχανισμούς που έχουμε στην βοήθεια που δίνει η Κομισιόν και διαχειρίζεται η Κομισιόν. Πρόσφατα οργανώσαμε μάλιστα ένα σεμινάριο για να δούμε τι συνέχεια θα δοθεί στις κατευθύνες γραμμές με τους συναδέλφους εντός της Επιτροπής, όπου είχαμε προσκαλέσει και την κοινότητα των ΜΚΟ. Να πω τέλος δύο λόγια για την έρευνα και την ανάπτυξη όσον αφορά τις τεχνολογίες αποναρκοθέτησης, που νομίζω είναι ένας τομέας ο οποίος δεν συζητάται επαρκώς. Well, just to highlight that I think from... Από την άποψη της Ένωσης και της Κομισιόν, εξ αρχής υποστηρίξαμε στεναρά την σύμβαση της ΟΤΑΒΑ, που όπως υπόθηκε ήταν μια μοναδική συμφωνία, ένα μοναδικό μέσο για τον αφοπλισμό όταν υιοθετήθηκε πριν από 10 χρόνια περίπου. Όταν μιλάμε για δράσεις για τις συνάρκες, βεβαίως δεν πρόκειται μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με αυτήν την υπόθεση και θέλω να υπογραμμίσω πως όλα τα κρατημέλη, τουλάχιστον αυτά που έχουν συνυπογράψει τη σύμβαση, 25 δηλαδή εκ των 27, Πολωνία και Φιλανδία δεν έχουν υπογράψει αυτό το μέσο, αλλά προγραμματίζουν να τον υπογράψουν μέχρι το 2012. Όπω σα είπα υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία κάνει η κοινότητα αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα κράτη-μέλη, διμερή δηλαδή βοήθεια. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το Συμβούλιο που μέσω του προπολογισμού ΚΕΠΑ έχει κάποιες ε, κοινέ δράσεις ε, όσον αφορά την υποστήριξη της παγκόσμιας αποδοχής της Σύμβασης της Όταβα και Όπως ε, ήδη υπόθηκε, όταν ε, κανείς εξετάζει τις δράσεις για τις νάρκες, βλέπει διάφορες δράσεις. Διάφορες δραστηριότητες οι οποίες ε, αναφέρονται εδώ, έχουμε την ίδια την αποναρκοθέτηση, την εκπαιδεία, την εξουδετέρωση των ε, αποθηκευμένων ναρκών. Αυτό είναι υποχρέωσή μας υπό την σύμβαση της ΟΤΑΒΑ. Επίσης ενημέρωση για τις νάρκες και βοήθεια φυσικά στα θύματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποστηρίξει 45 διαφορετικές χώρες ολόκληρο το κόσμο και κατά την περίοδο 2002 μέχρι 2008 έχουμε δαπανίσει γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ βλέπετε την κατανομή των αριθμών για τα περασμένα 6 χρόνια. Αλλά θέλω επίσης να προσθέσω ότι όταν βλέπουμε αυτή τη διαφάνεια, για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη ισχύω της σύμβασης της ΟΤΑΒΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει συνολικά 1,5 δις ευρώ σε δραστηριότητες κατά των αρκών. Αναμένοντα την επόμενη διαφάνεια, σα λέω ότι 500 από αυτά τα εκατομμύρια ήρθαν από κοινοτικού πόρου, μεταξύ των οποίων, όπω είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια, 300 εκατομμύρια δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 ετών. Έχει λεχθεί ήδη ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια δράση που να συνδυάζει την πτυχή της ασφάλειας και την πτυχή της αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν είναι ο κατάλληλος χώρος και χρόνος να συζητήσουμε το θέμα αυτό, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα γνωστό και είναι ίσως και στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Δεν μπορώ όμως να παραλείψω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι θεωρώ μερικές φορές ότι υπάρχει μια ανησυχητική τάση να προσπαθήσει κανείς να στρέψει τους δείκτες του ορολογίου προς την φορά αντίθετη αυτή των δικτών του ορολογίου σε ό,τι αφορά την πολιτική ασφάλειας που έχει ήδη προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γίνεται μια προσπάθεια να χωριστεί το τμήμα το οποίο αφορά στην ασφάλεια από το τμήμα που αφορά την άμυνα. Αυτό φυσικά είναι αποκοίημα της πυλωνικής δομής που έχουμε ακόμα μέχρι την έγκριση της, ε, της συνθήκης της Λισαβόνας. Καλό θα ήταν όμως να επιστηθεί η προσοχή της Επιτροπής σας στο σημαντικό αυτό γεγονός, το οποίο ενίοτε αποτελεί εγγενή αντίφαση στο συνολικό και οικουμενικό πλαίσιο αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών, διότι η δράση κατά των αρκών αποτελεί ένα εξέχον παράδειγμα αυτής της ε, κομβικής διασύνδεσης αναπτυξιακής βοήθειας και ασφάλειας, τώρα που έχουμε τις λεγόμενες κυρίου ρεύματο πολιτικές, mainstreaming δηλαδή, για την αντιμετώπιση των αρκών σε ένα αριθμό γεωγραφικών εργαλείων στη διάθεσή μας, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα την κομβική σύνδεση και διαπλοκή όλων αυτών των στοιχείων. Ήδη έγινε μνήα του γεγονότος ότι εδώ και δύο χρόνια δεν έχουμε πια μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού. Απλώς έχουμε κάποιες ε, γραμμές όπου περιλαμβάνεται και η εφαρμογή των διαφόρων γεωγραφικού χαρακτήρα εργαλείων. Πρέπει όμως να σας υπενθυμίσω ότι το γεγονός ότι οι ειδικά αφιερωμένες γραμμές του προϋπολογισμού καταργήθηκαν πριν από μερικά χρόνια. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας συνολικής μεταρρύθμισης μέσα στην οποία πολλές θεματικές γραμμές του προϋπολογισμού όπως παραδείγματος χάρη η αντιμετώπιση των ναρκωτικών και αυτή καταργήθηκε. Επομένως δεν είναι μια απόφαση η οποία εστρέφεται συγκεκριμένα κατά της αντιμετωπίσεως των ναρκών των δράσεων αυτών που ήταν αν θέλετε μια παράπλευρος απώλεια αυτής της μεταρρύθμισης. Μειώθηκαν τα εργαλεία από 40 σε 11 και αυτά τα 11 εργαλεία, τα 11 κύρια εργαλεία έχουν όλα τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τη δράση κατά των αρκών. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει μειωθεί η χρηματοδότηση, αλλά επειδή δεν υπάρχει πια η ειδική γραμμή του προϋπολογισμού μετά από το 2007, έχουμε ατενίσει μια κάποια μείωση των χρηματοδοτήσεων. Αξίζει όμως να εστιάσετε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ακόμα και όταν είχαμε μια αφοσιωμένη γραμμή του προϋπολογισμού, τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης των δράσεων κατά των αρκών ερχόντουσαν από γεωγραφικού χαρακτήρα γραμμές του προϋπολογισμού και μόνο ένα τρίτο από την τόσο αφιερωμένη και αφοσιωμένη αυτή γραμμή. Πρέπει επίση να υπενθυμίσω στους συναδέλφους μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα κατά γεωγραφικό χώρο εργαλεία το πόσο μεγάλη σημασία την οποία εμεί αποδίδουμε στην συνέχιση και την παρακολούθηση τη σύμβαση τη Οτάβα. Όχι αυτή καθεαυτή τη σύμβαση τη Οτάβα, αλλά των βασάνων τα οποία προκύπτουν όχι από τη σύμβαση τη Οτάβα, αλλά από τη μη καταστροφή των προστασίων και την πιθανή και ενδεχόμενη έκρηξη ναρκών. Αυτό έχει συμβεί λοιπόν στο παρελθόν και έχουμε ξεκινήσει και μια εξωτερική εκστρατεία για να γίνει γνωστό σε όλους τους συναδέλφους μας και στις Βρυξέλλες, στο αρχηγείο της Κομισιόν, αλλά και στα εθνικά κράτη, τις σημασίες που έχει ο εντοπισμός και η εφαρμογή των σχεδίων που λαμβάνουν χώρα Επιτοπίω, Ο κ. Χέρμπε αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πολλές φορές είναι πεπλεγμένο για αυτούς οι οποίοι είναι εκτός του νυμφώνος τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις συγκεκριμένα και άλλους να κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω απόλυτη κατανόηση γι' αυτό γιατί ούτε και εγώ τις καταλαβαίνω αυτές τις διαδικασίες τουλάχιστον δεν τις καταλάβαινα προτού γίνω μέλος της, ε, όταν έλθω να δουλέψω στην Κομισιόν. Αλλά οι κατευθυντήρε γραμμέ, τα δημόσια έγγραφα τα οποία έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο και υπάρχουν πολλά αντίγραφα πάνω στο τραπέζι, αυτά τα οποία περιλαμβάνουν το ότι όταν ξεκινάμε να αναπτύξουμε μια στρατηγική κατά χώρας, μια περιφερειακή στρατηγική επίσης, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να βασιστούμε σε ένα γενικό κατάλογο προτεραιοτήτων, ο οποίος να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση κατά των αρκών και επίσης υπάρχουν τα λεγόμενα ενδεικτικά προγράμματα και πολυετής δράσεις που καθορίζουν πιο συγκεκριμένα ποιες στρατηγικές θα ακολουθηθούν και είναι σημαντικό οι δράσεις κατά των αρκών να παραμείνουν σε ένα υψηλό σκαλί της κλίμακος προτεραιότητων. Αυτά τα ενδεικτικά προγράμματα αποτελούν αντικείμενο διαλόγου και διαπραγματεύσεων ενίοτε με τις χώρες αποδέκτριες. Επομένως, εναπόκειται και στις τελευταίες αυτές αποδέκτριες χώρες οι οποίες είναι και οι εποφελούμενοι και ευεργετούμενοι να καθορίσουν τις προτεραιότητες γιατί εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την αρρωγή προς μια χώρα όπως η Λευκορωσία ή η Ουκρανία όπως εδώ εδώ πέρα εφόσον αυτές δεν το επιθυμούν. Δίνουμε όμως μεγάλη σημασία στο να δώσουμε αρρωγή προς τις χώρες αυτές, ιδίως για να καταστρέψουν το υπολοιπόμενο οπλοστάσιο τους, ως ελέγχθη όμως αυτό είναι μία μάκρα και εσπαρμένη με άκανθες οδούς. Οδός. Υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα τα οποία παραμένουν και εξάλλου οι νάρκες της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας είναι ιδιαίτερα εξελιγμένες και εκλείουν ένα θανατηφόρο αέριο. Επομένως χρειάζεται ειδικό εξοπλισμός για τη διαδικασία καταστροφής τους. Έχει γίνει ένας δημόσιος διαγωνισμός Χρησιμοποιώντα αυτή την αφοσιωμένη γραμμή η οποία παρά την αφοσίωσή τη δεν υπάρχει πλέον. Και πολλές φορές οι διαδικασίες αυτές διαγωνισμού δεν ήταν επιτυχής. Γι' αυτό έχουμε ενθαρρύνει την Ουκρανία και τη Λευκορωσία να θέσουν υψηλά στον κατάλογο προτεραιότητών τους την καταστροφή αυτού του οπλοστασίου. Και ελπίζω λοιπόν ότι ακολουθούμε την, την ορθή κατεύθυνση ήδη στην ε, Λευκορωσία και προσεχώς και στην Ουκρανία. Αυτό θα σημαίνει ότι στην Καρθαχένη των Ινδιών ή μάλλον της Κολομβίας η Ουκρανία θα ανακοινώσει ότι μπορεί να καταστρέψει και τις ε, υπόλοιπες νάρκες της μέσα σε ένα ορατό μέλλον. Δεν χρειάζεται βέβαια να υπενθυμίσω την Επιτροπή σας ότι τίθεται και θέμα πολιτικής θέλησης και ιδιαίτερα για την Ουκρανία αυτό έχει αντιμετωπιστεί και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Προέδρου της ε, Επιτροπής και της Πρωθυπουργού της κυρίας Τιμοσέγκο. Ίσως επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα να τονίσω ότι είχαμε οργανώσει ένα σεμινάριο για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ξεκίνησε ως πρόγραμμα εκπαίδευσης και είχαμε προσκαλέσει και τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ένα τμήμα αυτού του σεμιναρίου εστόχευε ήταν για να υπενθυμίσει στους συναδέλφους μας και να τους εξηγήσει ποιες είναι οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό και επίσης να τους ε, υπενθυμίσει την ύπαρξη μιας ενδιάμεσης αναθεώρησης για πολλά προγράμματα και εργαλεία που αποτελεί εξάλλου και μια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε τις νέες εξελίξεις ακόμα και τη σημασία που αποδίδουμε στη δράση κατά των ναρκών. Εν τέλει, είχα υποσχεθεί να σας πω και μερικά λόγια για την έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα αυτό. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είμαι η για τα θέματα αυτά. Οι συνάδελφοί μου από την Γενική Διεύθυνση του Επιχειρήν είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά έρευνας και ίσως αν ήταν εδώ σήμερα θα μπορούσαν να σας εξηγήσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ απλώς υπογραμμίζω το γεγονός ότι εμείς υποστηρίζουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα αυτό σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες ναρκοθέτησης και υπάρχει ένα σημαντικός προϋπολογισμός ο οποίος είναι διαθέσιμος <clears throat> στον τομέα αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για έρευνα ασφαλείας που κυρίως αφορά την, ε, τα θέματα ασφαλείας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς να αντιμετωπίζουμε και να εντοπίζουμε τα εκρηκτικά είναι 1350 ευρώ είναι μάλλον 350 εκατομμύρια ευρώ σε επταετή περίοδο, εμείς εξασφαλίσουμε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των κονδυλίων πηγαίνει για, την, για τον εντοπισμό και την ανείχνευση των αρκών. Και σας ευχαριστώ. Thanks very much. And now my colleague, Mr. Van Orden. Uh, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που έχουμε σήμερα εδώ από το Διεθνές Κέντρο της Γενέβης και ιδιαίτερα από τον Ερυθρό Σταυρό. Και θέλω ιδιαίτερα να τιμήσω τον Πίτερ Χάρμπι που τα τελευταία 20 χρόνια περίπου έχει ταχθεί, ταχθεί σε αυτό το σκοπό και εξακολουθεί να προσπαθεί. Και οι συνάδελφοί σα βέβαια δεν είναι όλοι εδώ σήμερα, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στι ε, δράσεις για τι συνάρκε, ε, αλλά βλέπουμε με θετικό τρόπο και τη συμβολή της ίδια της Κομισιόν. Ε, και νωρίτερα έχει, έχει γίνει πρόγραμμα και στο κοινό ερευνητικό πρόγραμμα κέντρο μάλλον. Από τεχνολογική άποψη υπήρξαν λοιπόν θετικές συμβολές εγώ συμμετείχα στην ε, ε, συμμετείχα στην προσπάθεια να γίνει τελικά η σύμβαση αυτή αρχικά από την, στην πόλη του Καναδά την οποία εγώ επισκέφθηκα πολλές φορές από το 1996 μέχρι το 1998 και κατάληξα να την γνωρίζω πολύ καλά ε, και υποστήριξα χορηγώντας ε, την αποναρκοθέτηση, την εξουδετέρωση ναρκών και την, κάλυψη, την ε, περίθαλψη των θυμάτων. Ορισμένοι από εμά ελπίζαμε ότι δεν θα διαρκούσε για πάντα αυτή η ενασχόληση με τις, με τις νάρκες. Μάλιστα είχαμε σκοπεύσει αρχικά να εξαλείψουμε αυτή την πληγή, την μάστιγα των ναρκών στα επόμενα δέκα χρόνια. Αλλά όπως βλέπουμε Ακόμα με αυτό ασχολούμαστε. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος βέβαια, τα ακούσατε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. 156 κράτη έχουν συνυπογράψει την συνθήκη της Όταβα, τεράστιες περιοχές έχουν καθαριστεί και έχουν, ε, καταστεί, έχουν, ε, έχουν ε, χαρακτηριστεί ελεύθερες ναρκών, έχει μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων, από Νάρκε, αλλά παρόλα αυτά έχει πρόσφατη καταμέτρηση 5.500 κόσμος, 5.500 ήταν τα θύματα από τι νάρκε κατά προσωπικού και άλλων εκρηκτικών ε, καταλήπων πολέμων. Πολλά έχουν αλλάξει λοιπόν, αλλά κατά κάποιο τρόπο και πολλά έχουν μείνει τα ίδια και παράλλαχτα. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος, αλλά μας έχει πάρει χρόνο να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα και υπάρχουν και βέβαια συγκεκριμένα συμφέροντα σε αυτήν την ε, συνεχιζόμενη υπόθεση με την οποία ασχολούμαστε όλοι. Από το 1967 η διεθνή κοινότητα έχει δαπανίσει περίπου 4 δις δολάρια σε δράσεις κατά των αρκών και εξακολουθεί να δαπανά μισό δις δολάρια ετησίως. Πολλά χρήματα, πολλά χρήματα δαπανώνται για αυτή την υπόθεση. Κατά την έποψή μου, θα πρέπει, θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο και να φτάσουμε σε ένα τέλος μόνο όμως αυτό μπορεί να γίνει αν επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες ε, τρεις πτυχές. Καταρχήν το πολιτικό ζήτημα. Εδώ και χρόνια έχει υπάρξει πολύ μεγάλη ε, αντιπερισπασμό σε σχέση με το πολιτικό θέμα. Δηλαδή, η πολιτική μας εκστρατεία θα πρέπει να απευθύνεται όχι στα, στις ΙΠΑ, που ήταν ε, ο στόχος, κατεξοχήν στόχος τα πρώτα χρόνια, λόγω των δικών τους πολιτικών κινήτρων. Μάλιστα, οι ΗΠΑ έχουν συμβάλει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη χώρα στο θέμα, στην υπόθεση της απονορκοθέτησης και εξακολουθεί να ισχύει αυτό. Το 2007 έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθησε η Νορβηγία 50 εκατομμύρια, Καναδά 46, έπειτα η Κομισιόν με 45 εκατομμύρια και από τα κράτη-μέλη της Ένωσης το Ηνωμένο Βασίλειο και οι κάτω χώρε είναι πάνω-πάνω στη λίστα. Δίνουν, έδωσαν περίπου 25 εκατομμύρια το χρόνο. Η Γερμανία και η Σουηδία ακολουθούν κατά πόδας. Και η Γαλλία δυστυχώς εδώ έχει ε, κάνει την εξαίρεση. Εδώ έχει συμβάλει πολύ λίγα, με ένα μέσο όρο 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Η πραγματική ένοχη που ανέφερα λοιπόν είναι οι χώρες αυτές που εξακολουθούν να παράγουν νάρκες κατά προσωπικού και να τις εξάγουν κιόλα. Όσον αφορά τους παραγωγούς βέβαια, η Κίνα, η Κούβα, το Ιράν, η Βυρμανία, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και ένα δυο άλλοι. Ορισμένες από αυτές τις χώρες, η Κίνα και η Ρωσία αναφέρθηκαν έχουν ε, εφαρμόσει απαγόρευση εξαγωγών εδώ και χρόνια, αλλά το Ιράν, ας πούμε, ισχυρίζεται ότι έχει σταματήσει τις εξαγωγές, ενώ υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο. Αλλά βέβαια, μεγαλύτερη ένοχη είναι αυτοί που εξακολουθούν να δημιουργούν τον θάνατο μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης των αναρκών κατά προσωπικού, όχι οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις βέβαια, που είναι υπεύθυνε δεν ε, κάνουν πόλεμο αδιακρίτως, αλλά οι Ρώσοι, οι Βερμανοί, οι Βερμανικοί στρατοί και οι Ρωσικοί στρατοί χρησιμοποιούν τους νάρκες, δημιουργούν ε, θύματα, προκαλούν θύματα και πιο σημαντικό είναι οι μη κρατικέ ένοπλες ε, ομάδες για να χρησιμοποιήσουμε το πιο ευγενικό όρο, δηλαδή τους, ε, ε, τους ε, ταραξίες και τους τρομοκράτες. Αυτές οι ομάδες είναι που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον αθώο άμαχο πληθυσμό, καθώς και στις νόμιμες ένοπλες δυνάμεις. Οι κύριοι καταχραστές, και θα πρέπει αυτό να το διαβάσουμε από το Landmine Monitor, που σας το συστήνω την έκθεση αυτή μάλιστα να τη διαβάσετε, είναι μια εξαίρετη δημοσίευση. Οι κύριοι καταχραστές είναι η, τα Mill Tigers, η ATT στη Σρι Λάγκα, μεγάλος χρήστης και καταχραστής αυτών των ε, ναρκών ε, αντιπρο, κατά προσωπικού είναι η ΦΑΡΚ στην Κολομβία, η Ταλιμπάν και ένα σωρό άλλοι τέτοιοι που είναι η πραγματική ένοχη και καταχρώνται των ε, ναρκών. Οι προσπάθειές μας θα πρέπει επίσης να επιστιαστούν σε συγκεκριμένες, ε, ε, συγκεκριμένους τομείς. Πολλοί πόροι και προσπάθειες έχουν δαπανηθεί σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν ενάρκες. Το ξέρουμε το πρόβλημα αυτό εδώ και μια δεκαετία ή και παραπάνω. Είναι η αντίληψη του κινδύνου που κυριαρχεί στις δραστηριότητές μας πάνω από μια δεκαετία μετά τη συνυπογραφή της συνθήκης για την απαγόρευση των ναρκών, μια πραγματική αξιολόγηση αξιόπιστη εξακολουθεί να μην υπάρχει. Και αυτό σας το αναφέρω από το Landmine Monitor. Λιγότερο από το 3% της γης που έχει καθαριστεί, καθαριστεί περιείχε πραγματικά νάρκες ή άλλους συγκριτικούς μηχανισμούς. Αναφερθήκατε στις αρχές της απελευθέρωσης της ε, γης, δηλαδή πρώην ύποπτες περιοχές σε μεγάλες ε, ε, επιφάνειες απελευθερώνονται για χρήση χωρίς να περνάμε από δαπανηρώσεις και χρονοβόρες προσπάθειες για καθάριση από τη στιγμή που δεν χρειάζεται καθάριση. Εγώ κατανοώ τα προβλήματα όσον αφορά την πραγματική εξακρίβωση, εξακρίβωση της ασφάλειας αυτών των περιοχών, για να μπορεί δηλαδή ο κόσμος συνεχίσει να ζει εκεί. Αλλά σαφώς πλέον επιτέλους υπάρχουν τρόποι για να ξεπεράσουμε ένα τμήμα αυτού του προβλήματος. Να σας πω πως ε, σε αυτό το πλαίσιο εκείνοι που ξεπερνούν μάλλον από την σύμβαση της ΟΤΑΒΑ αναλαμβάνουν πολύ σοβαρές υποχρεώσεις. Μία από αυτές είναι ότι πρέπει να καθαρίσουν επικράτεια που είναι υπό τον έλεγχό τους. Να αναφέρω ένα παράδειγμα των νήσων Φόκλαντ, γιατί όταν το Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνει στο εδόλιο του κατηγορουμένου επειδή δεν έχει συμμορφωθεί με την σύμβαση της Οτάβα είναι γιατί δεν έχει καθαρίσει τα νησιά Φόλκλαντ, την ίσο Φόλκλαντ. Και δεν το έκανε γιατί δεν είχε χρήματα. Είναι, ε, μάλλον, είναι χρήματα και χρόνος όμως που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ καλύτερα σε άλλα μέρη. Μιλούσαμε εκπροσώπους από τα νησιά Φόκλαντ, στο Μάντσεστερ, στην... την περασμένη εβδομάδα σε μια συνεδρίαση και έλεγαν πως είναι απόλυτη... ήταν απόλυτη ανοησία. Γιατί όποιος γνωρίζει τα νησιά και εγώ έχω πάει εκεί, είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή κατοικείται από καμιά εκατοστή ανθρώπου και γύρω στα 2 εκατομμύρια πρόβατα. Πολύ όμορφη περιοχή. Υπάρχουν μεγάλε εκτάσει που υπάρχουν υποψίε για νάρκε κατά προσωπικού που βασικά έβαλαν οι Αργεντινοί όταν ε, εισέβαλαν στα νησιά Φόλκλαντ. Εξακολουθεί να είναι εκεί, αλλά δεν βλάπτουν κανέναν. Η προσπάθεια που απαιτείται για την καθαρισμό αυτών των περιοχών είναι τεράστια, είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Και τα χρόνος και το χρήμα θα μπορούσαν πιο επωφελώς να χρησιμοποιηθούν άλλου. Το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω είναι η χρήση των ενόπλων δυνάμεων. Το τμήμα του κόστους της χρήσης ε, πόρων ε, από τις ε, ένοπλες δυνάμεις ή από το πολιτικό προσωπικό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κανένας υπολογισμός. Ανέκαθεν εγώ θεωρούσα ότι σε ε, χώρες όπου είχαν ένοπλες σειράξεις, οι πρώτοι που θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους είναι οι ένοπλες δυνάμεις για να καθαρίσουν. Μιλώ κυρίως για τη Βοσνία. Διότι το πρόβλημα αυτό διονύζεται στη Βοσνία. Και επίσης θα έλεγα ότι η κατάσταση εκεί είναι ε, απαράδεκτη τελείως. Είναι πολύ αργοί οι ρυθμοί καθάρισης. Υπάρχουν ακόμα ατυχήματα στην αποναρκοθέτηση και θύματα απονάρκες εξακολουθούν να πέφτουν. Είναι ένα ε, συνεχές και συνεχιζόμενο πρόβλημα και εκεί υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να καταρτιστούν, να αναπτυχθούν για να συμμετέχουν περισσότερα στην αποναρκοθέτηση στη Βοσνία. Με εκπλήσει πάρα πολύ γιατί δεν κάνουμε μεγαλύτερη πρόοδο εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, μερικά σημεία ακόμα για την τεχνολογία. Και βέβαια, με την πάροδο των ετών, όλοι αγωνιστήκαμε σκληρά για να προσπαθήσουμε να βρούμε νέες τεχνολογίες για να εφαρμοστούν σε αυτό το πρόβλημα. Και θυμάμαι πριν από πολλά ε, χρόνια ε, πολλές ιδέες, πολύ ευρηματικές και πολύ εφάνταστες δεν ξέρω, γάτες, σκυλιά, από ένα αέρια μέσα, ακούστηκαν διάφορα. Και διάφοροι τύποι ε, εκεί εμφανίζονταν με την τελευταία ιδέα που τους είχε κατεβεί. Πάντως, έχουμε, επαναλαμβάνω, ένοπλες δυνάμεις που ασχολούνται και ανισχούν ε, με τις απειλές με, ε, τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί. Εκπλήσωμε. Γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. ή με αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, α πούμε. Ε, υπάρχει αυτό ο προβληματισμός στην ε, και στι ένοπλες δυνάμεις. Έχουν λοιπόν μεγάλε προόδοι και τεχνολογικά, ωστόσο θα πρέπει να θέσουμε νέες προτεραιότητες. Βεβαίω θα συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εσωτερικό μας, αλλά χρειάζεται και μεγαλύτερη εστίαση. Απογοητεύομαι που μετά από όλα αυτά τα χρόνια που θεωρούσαμε ότι θα έχουμε και αγωνιστήκαμε για να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση και ένα νέο κονδύλι, μια θέση στον προπολογισμό, γιατί υπήρχαν εσωτερικοί συσχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαμάχες που καταλαβαίνουμε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ε, και είχαμε κάπως χαλαρώσει μετά από αυτή την προσπάθεια. Είναι κρίμα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει και ε, με χρηματοδότηση βέβαια ενημιούμενη αυτή ε, γενικά συμφωνώ πάρα πολύ με την περικοπή των κοινοτικών κονδυλίων αλλά για το συγκεκριμένο ε, Ακριβώ υπό την προπόθεση να χρησιμοποιούνται καλά τα κονδύλια και να πηγαίνουν σε σωστή κατεύθυνση, είμαι υπέρ τη διατήρηση τη μεγάλη χρηματοδότηση. Ένα τελευταίο, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στι ανάγκε των θυμάτων. Διότι σε τελική ανάλυση Περί αυτών πρόκειται. Θέλουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, να βελτιώσουμε την ευκαιρία που έχουν οι συνάνθρωποι μας στη ζωή και να τους ε, ελαφρώσουμε κάπως, να ε, καταπραίνουμε ε, αυτή τη, τον πόνο και τα δεινά που ζουν. Είναι πολύ σκληρή πραγματικότητα. Όταν κάποιος χάνει ένα πόδι και τα δύο ή ένα χέρι και τα δύο είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον τόσο δύσκολο. Και αυτό ε, χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. you very much, Mr. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φανόρντεν. Και τώρα κυρία Μπάτνερ που είναι η συγγήτρια του εργαλείου σταθερότητος. Ευχαριστώ μου δίνετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετέσχουν σε αυτό το σεμινάριο. Ευχαριστώ και το Τμήμα Πολιτικής για την διοργάνωση αυτή. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή που μπορούμε να κάτσουμε και να σκεφτούμε για αυτό το θέμα που είναι θέμα ανθρώπινης ασφάλειας. Μιλήσατε για την πτυχή της ασφάλειας, την πτυχή ανάπτυξης. Για μένα όμως ο τρόπος προσέγγισης σε αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι η ανθρώπινη ασφάλεια. Έτσι πρέπει να το ατενίσουμε το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπογραμμίσω ότι και η Κομισιόν το έθεσε αυτό το θέμα επιτάπητος λέγοντας ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτό το στοιχείο από τις θεσμικές μάχες οι οποίες μένονται. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει <clears throat> και η νέα υπηρεσία διεθνών, διεθνούς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το ζήτημα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να ευνοήσουμε ακόμα περισσότερο την ανθρώπινη ασφάλεια. Δεν πρέπει να το χάσουμε από τον βλεφάρων μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να, θέσει, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να τονιστεί και αυτή η πτυχή του προβλήματος. Η σύμβαση της ΟΤΑΒΑΣ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί από τους υπέρμαχους δράσεις από την κοινωνία των πολιτών στον τομέα αυτό και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υποφελώς αυτό το παράδειγμα και αλλού. Εγώ, σαν εισηγήτρια για το μέσο σταθερότητα, θα ήθελα να έχω κάποιες διαβεβαιώσεις από την Κομισιόν για το πώς θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα πιο θετικό μήνυμα στην Σύνοδο της Καρθαγέννη, γιατί το θέμα αυτό παραμένει εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ελέγχθη <clears throat> προηγουμένως, υπήρχε μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού, η οποία τώρα έχει αντικατασταθεί από μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών. Θα ήθελα να ξέρω από την Κομισιόν ποια είναι τα στοιχεία που έχετε ότι οι κατευθυντήριες γραμμέ σα για την ενσωμάτωση σε όλε τι πολιτικέ της δράση κατά των ναρκών θα είναι μια υποφελή αντιμετώπιση. Και τι έχει να πει το αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι υπήρξε πραγματικά μείωση της χρηματοδότησης κατά των αρκών και πώς θα επιτύχετε το στόχο του να διατηρήσετε ένα υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης στον τομέα αυτό. Επίσης και πάλι από την οπτική γωνία του μέσου σταθερότητος πώς θα ε, διευρύνετε τις δράσεις κατά των αρκών μέσα στα πλαίσια του μέσου σταθεροποίησης. Και επίσης στην Καρφαγέννη πώς θα μπορέσετε να αυξήσετε το προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας κύριας δύναμης που θέλει να παίξει ρόλο στον τομέα της αποναρκοθέτησης. Επίσης, μετά από την Καθαγέννη και στην επόμενη, εν ώψη της επόμενης διάσκεψης του 2014, τι θα πράξει η Κομισιόν μέχρι τότε. Θέλω επίση να στραφώ και προς το Συμβούλιο και να ξέρω ποια είναι η θέση που θα αναλάβει το Συμβούλιο στην Καθαγέννη για να διευρύνει την ε, εμβέλεια των ε, ναρκών που καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα, όχι δηλαδή μονάχα τι νάρκες προσωπικό, αλλά και τι νάρκες κατά οχημάτων και αρμάτων. Τώρα, για τι βόμβε διασπορά, για του οπλισμού διασπορά που δεν θα αντιμετωπιστούν στην Καρθαγέννη. Δεν φαίνεται όλα τα κράτη-μέλη να επιτυγχάνουν το στόχο τους μείωσης ή καταστροφής των αποθεμάτων τους για αυτούς τους οπλισμούς. Θα ήθελα να ξέρω τι κάνει η Σουηδική Προεδρία σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Έχουμε καθυστερήσει μισή ώρα, λέει ο Προεδρεύων, και αρχίζουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κυρία Μπράτνερ. Ποιος θα ήθελε να λάβει τον λόγο τώρα. Ο κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ. Μόλις γύρισα από την Αντίσα Μπέμπα, όπου συζητείται η εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Αφρικής. Και ετέθη το ερώτημα, πώς συναρμόζεται αυτή η δραστηριότητα της αποναρκοθέτησης στη στρατηγική μας έναντι της Αφρικής. Υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο το οποίο έχει συμφωνηθεί για τη δράση μας στην Αφρική. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. But... Ευχαριστώ. Ο, κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη απευθύνεται στο ε, Διεθνές Κέντρο της Γενέβης. Είπατε ότι για μια πιο συνεκτική και στρατηγική προσέγγιση, λέτε, χρειάζεται μεγαλύτερη πραγματογνωμοσύνη αλλά και χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να μας το συγκεκριμενοποιήσετε λίγο αυτό, για να διευκρινιστεί ακριβώς τι σημαίνει αυτό στην πράξη κατά την άποψή σας. Η δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Χέρμπι. Τονίσατε την ανάγκη να παραμείνουμε σε μια νοοτροπία κουλτούρα συμμόρφωσης και τήρησης των κανόνων. Θέλετε και μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποια είναι τα σημαντικότερα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Και τρίτη ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Σουηδικής Προεδρίας. Η Ελλάδα, είπατε, είναι μία από τις χώρες που με επανειλημμένα στη συζήτηση και ακούσαμε και σήμερα ως χώρα που αθετεί την υποχρέωσή της για καταστροφή των αποθεμάτων. Ε, ποια βήματα προτείνετε εσείς και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να κινηθεί η Ελλάδα προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης. Ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε, εξέχοντα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριοι συνάδελφοι, ονομάζομαι Λιδία Πνευματικού, είμαι νομικός σύμβουλος στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στις Βρυξέλλες και είμαι επιφορτισμένη να παρακολουθώ την ομάδα για τον παγκόσμιο εφοπλισμό κοντούν του Συμβουλίου. Ε, επειδή στην σημερινή μας συζήτηση η Ελλάδα αναφέρθηκε πολλές φορές ως κράτος το οποίο δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τη Σύμβαση της Οτάβας, θα ήθελα μόνο να πω δύο λόγια εξ όσων γνωρίζω ε, για την πρόοδο της καταστροφής των ναρκών από τη χώρα μας. Ε, η Ελλάδα έχει ήδη καταστρέψει 33% από τα αποθέματά της. Ελπίζει ότι το 50% των αποθεμάτων θα έχουν καταστραφεί πριν από τη Σύμβαση της Καρθαγένης, ώστε να μπορέσει να το ανακοινώσει εκεί. Ε, επίσης πρέπει να πω ότι επειδή υπάρχει μεγάλη δυσκολία ως αδυναμία να καταστραφούν οι νάρκες στο ελληνικό έδαφος, έχει γίνει συμφωνία με τη Βουλγαρία και οι νάρκες ε, μεταφέρονται στη χώρα αυτή, η οποία έχει τα μέσα για την καταστροφή τους. Ε, και η Ελλάδα διαθέτει επίσης τα πρωτόκολλα καταστροφής των ναρκών που έχουν ήδη καταστραφεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έγινε ερώτηση για την πραγματογνωμοσύνη και τη χρηματοδότηση. Και τι εννοούμε. Αν μου επιτρέπετε να σας πω μόνο ότι αυτό το θέμα της γεωγραφικής μετατόπισης δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κέντρο της Γενέβης για τις Νάρκες. Ε, είπαμε ότι δίνονται χρήματα για την έρευνα, για την τεχνολογία. Αυτά τα αναλαμβάνει η στρατιωτική βιομηχανία. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πρόκειται για στρατηγικό ανασχεδιασμό για τη χρήση των γεών που απελευθερώνονται, δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση αλλά στο στάδιο της εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων τελικά θα έχουμε εξοικονόμηση πόρων. Δεν είναι δαπανηρό αυτό. Υπάρχει δυσκολία στην ε, καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτής της αντίληψης. Θα σας ε, δώσω τώρα το λόγο κύριε Πάτερσον, γιατί ο κύριος ε, Πάτερσον έχει κάνει τη μελέτη. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση λείπουν και κονδύλια και εμπειρογνωμοσύνη. Εδώ μιλούμε για κονδύλια που έχουν χαθεί ε, και ελέγχονται από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κεντρικά στις Βρυξέλλες και περιορίζεται και ε, η θέση στον προπολογισμό αλλά περιορίζεται σε στελέχωση και η μονάδα στη Ρέλεξ και σε κάποια άλλη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, έχει επικεντρωθεί εκεί. τα κονδύλια που υπάρχουν μπορούν να χρησιμοποιούν στρατηγικά ε, και ε, παγκόσμια πρόπτικη και υποστηρίζουμε και τις αντιπροσωπείες ε, για το σχεδιασμό και για τη δράση όταν πρόκειται για χάραξη προτεραιτήτων σε γεωγραφικό επίπεδο. Γι' αυτό μιλάμε συγκεκριμένα, δεν είναι γενικά ότι έχουμε πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω στο ένα ερώτημα το οποίο απευθυνόταν σε μένα σε σχέση με το πρόβλημα της συμμόρφωσης και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Η πρώτη ευκαιρία που έχουμε ενώπιόν μας είναι η διάσκεψη της Καρθαχένας, Καρθαχένης. Είναι απαραίτητο να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα, το οποίο να μην συγκαλύπτεται με διπλωματικούς όρους, αλλά να είναι σαφές προς όλα τα συμβαλόμενα κράτη-μέλη ιδίως για τον τομέα της ε, αποναρκοθέτησης και εκαθάρισης, για να τονίσουμε ότι η νομική υποχρέωση είναι να υπάρξει εκαθάριση το ταχύτερο δυνατόν και όλα τα κράτη τα οποία έχουν τέτοιες συμβατικές υποχρεώσεις και δεν τις έχουν εκπληρώσει ακόμα, θα πρέπει να θέσουν όλους τους απαραίτητους πόρους στην διάθεση της διαδικασίας εκαθάρισης αντιμετωπίσαμε προβλήματα γιατί όλοι περιμέναν μέχρι τον 8ο, 9ο ή ακόμα και 10ο χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης για να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή από αναρκοθέτηση και φυσικά αυτό δεν ήταν επαρκές. Επίσης για την καταστροφή των οπλοστασίων νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάσκεψη της Καρθαχένης να τονίσει προς τα συμβαλόμενα αυτά μέρη τα οποία δεν έχουν καλύψει ή δεν θα καλύψουν τις καταληκτικές προθεσμίες να του ζητήσει κατεπηγόντως <clears throat> να καταβάλουν προσπάθειες για τη συμμόρφωσή τους και να ανακοινώσουν τις καταληκτικές ημερομηνίε για το πρόγραμμά τους, αν δεν το έχουν πράξει ακόμα, τουλάχιστον το κάνουν στην Καρθαγέννη. Για την αρρωγή προς τα θύματα θα πρέπει και πάλι να υπάρχουν χρονικά δεσμευτικές ε, αναλήψεις υποχρεώσεων για την παροχή αρρωγής στα θύματα σε συγκεκριμένες περιοχές και επίσης και μια μεγαλύτερη εστίαση να αναλάβει το κάθε κράτος της την πρωτοβουλία για τι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, γιατί σε κάποια κράτη δεν είναι η προτεραιότητα, μπορεί η προτεραιότητα να είναι απλώ στην αντιμετώπιση των θυμάτων και όχι στην γενικότερη περίθαλψή του. Αν δεν υπάρξει λοιπόν εθνική πρωτοβουλία και ανάληψη ευθύνη για τα θέματα αυτά, δεν μπορούμε να πράξουμε τίποτα. Για το θέμα των διαθεσίμων πόρων, νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμεί σε πρακτικό επίπεδο να έχουμε μια μόνιμη επιτροπή η οποία θα αντιμετωπίζει το θέμα αυτό κάθε χρόνο σε μόνιμο επίπεδο, ώστε οι πληροφορίες από την Κομισιόν, από τα κράτη-μέλη, από τους δωρητέ, από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να συλλεγούν και να συνταρμοστούν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό εδώ να δούμε κατά πόσο η κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση μιας οικουμενικής δράσης και εφαρμογής στον τομέα των αρκών αν θα μπορέσει ποτέ να γίνει πλήρως πραγματικότητα μέσα στα πλαίσια των εργαλείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και κατά πόσο αυτά τα εργαλεία είναι επαρκή για την επίτευξη των προσδοκομένων στόχων. Διότι, για να είμαι ειλικρινής, σε μερικές από τις χώρες που πλήττονται από το πρόβλημα των αρκών υπάρχουν τόσες πολλές αντικρουόμενες προτεραιότητες που η εκαθάριση των αρκών ή η αρρωγή προς τα θύματα δεν θα είναι ποτέ μία από τις πρώτες προτεραιότητε. Αν έχετε χώρες που έχουν να αντιμετωπίσουν το AIDS, έχουν να αντιμετωπίσουν δεκάδες χιλιάδων θυμάτων από τροχαία ατύχηματα κάθε χρόνο, ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα σε αναπτυξιακό επίπεδο. Υπάρχουν και πολλοί, πολλές χώρες όπου η εκαθάριση των αρκών δεν λαμβάνει χώρα και ούτε καν θα τύχει δικαιολόγηση ως ανθρωπιστικός στόχος, παραγωγός χάρη, στα Falklands. Αν όμως παραμείνουν οι νάρκες σε μέρη όπου δεν απειλούν άμεσα τους άμαχους, τους πολίτες, θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση που το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις, ότι μένουν οι νάρκες ε, στο έδαφος και αυτό είναι σαν να χρησιμοποιούν νάρκες κατά προσωπικό. Ένα κράτος το οποίο έχει πάρει μια παράταση διατηρεί ακόμα χιλιές νάρκες γύρω από μια στρατιωτική βάση δεν τις έχει εκαθαρίσει, αυτό δεν είναι ανθρωπιστικό θέμα, αλλά αποτελεί συνέχιση της χρήσεως των ναρκών αυτών. Αυτό λοιπόν παραβιάζει τους στόχους της ε, σύμβασης και τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν δεν είναι μονάχα, οι στόχοι μας δεν είναι μονάχα το πλαίσιο ανάπτυξης, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα χρησιμοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το, ο κ. Μπούντικοφερ θέλει να θέσει άλλο ένα ερώτημα. Όχι, δεν θέλω να θέσω συμπληρωματικό ερώτημα θα ήθελα να αναθέσω στην ελληνική αντιπροσωπεία ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Και ο κύριος Φαν Όρντεν. Νομίζω ότι και ο, προ... ο εκπρόσωπος της Προεδρίας ήθελε να μου απαντήσει στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Η Προεδρία διατηρεί διμερείς επαφές με την Ελλάδα για το θέμα αυτό. Ακούσαμε την εξήγηση που έδωσε η Ελληνίδα μόνιμη αντιπρόσωπος εδώ και έχουμε εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι είναι ενεκτυλήξη μια διαδικασία και θα μπορέσει η Ελλάδα να ανακοινώσει μια καταστροφή του προστασίου κατά 50% όταν θα συναντηθούμε στην Καρθαγένη. Είναι λυπηρό όταν μια χώρα παραβιάζει τις συμβατικές της ε, υποχρεώσεις βάσει της ε, σύμβασης της ε, ΟΤΑΒΑΣ το ίδιο ισχύει και με την Τουρκία η οποία φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να καταστρέψει τις νάρκες της στο προσεχές μέλλον. Για τις άλλες ε, δύο χώρες που αναφέραμε, την ε, Λευκορωσία και την Ουκρανία, υπάρχουν ήδη διαδικασίες. Για τα δύο θέματα τώρα τα οποία τέθηκαν από την εισηγήτρια του Μέσου Σταθερότητος, θα ήθελα να σα ζητήσω να τι επαναλάβετε. Δεν είμαι σίγουρο ότι κατάλαβα πολύ καλά σε τι αναφέρεστε. Λυπάμαι αν δεν ήταν σαφές. Καταρχήν, το θέμα της ε, στάσης που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Καρθαγένη και το πόσο αυστηρή θα είναι αυτή η στάση, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν προσπάθειες να διευρυνθεί το αντικείμενο εκεί και να μην είναι μονάχα οι νάρκες κατά προσωπικό αλλά και οι νάρκες κατά οχημάτων. Σε ποιο βαθμό θα υπάρξει λοιπόν διεύρυνση του αντικειμένου και δεύτερον για το πλωστάσιο βοβών διασποράς στην Ευρώπη και κατά πόσο εσείς προχωρείτε να παροτρύνετε τα κρατημένα να καταστρέψουν ταχύτερα αυτό το απλοστάσιο. Για τα δύο αυτά θέματα δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφέρω γνώμη ως εκπρόσωπος της Προεδρίας. Αλλά αν θέλετε να ξαναγίνω Σουηδός, Μπορώ να σας πω ότι το θέμα άλλων ναρκών, όχι ναρκών κατά προσωπικού, αυτό αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια της σύμβασης για τα συμβατικά όπλα και αντιμετωπίζεται εδώ και αρκετά χρόνια, παραμένει ακόμα επιτάπητος και εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ανανεώσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν, γιατί τα πέντε αυτά χρόνια έγινε σημαντικό έργο στον τομέα αυτό των ναρκών. Δεν επέτυχαν, δεν ε, ευδοκίμησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις που ήταν πολύπλοκες και δύσκολες. Ελπίζουμε θα αναζωογονηθούν και θα ανανύψουν. Για τα όπλα διασποράς, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών και δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένε χώρες έχουν υπογράψει, όπως ξέρετε, την ε, σύμβαση της Οτάβας, αλλά κρατημέλη την έχουν υπογράψει. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε προς το παρόν τουλάχιστον είναι ένα πρωτόκολλο και πάλι μέσα μέσα στο, στη συζήτηση για τα συμβατικά όπλα που θα μπορέσουν να περιλάβουν και πρωτόκολλα τα οποία δεν θα απαγορεύσουν μεν αλλά θα ρυθμίσουν τη χρήση των όπλων διασποράς. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομος. Για τα ερωτήματα που ετέθηκαν για τις κατευθυντήριες γραμμές κατά των, τις δράσεις κατά των αρκών. Είναι ίσως πρόωρο το να αποφασίσουμε αν θα μπορέσει να αναχαιτιστεί η κατιούσα αυτή που έχει λάβει η πορεία της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ναρκών οι κατευθυντήρες γραμμές εγκρίθηκαν σαν έγγραφο εργασία της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης πριν από ένα χρόνο μονάχα περίπου. Ακολουθούμε λοιπόν, παρακολουθούμε μάλλον τι κάνουν οι γεωγραφικές μας μονάδες και αντιπροσωπείες και έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο των ε, εστιακών σημείων γιατί το θέμα δεν είναι μονάχα να έχουμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι δουλεύουν σε μία υπηρεσία της Κομισιόν. Είναι επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο να έχουμε τέτοιους εμπειρογνώμονες για την ε, αγροτική ανάπτυξη, την ε, ανθρωπιστική δράση, την ε, καθάριση των αρκοπεδίων. Γι' αυτό για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τις κατάλληλες στικές για το τι επιτυγχάνεται και υπάρχει πάντα κάποια καθυστέρηση μέχρι να μπορέσουμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχει δαπανηθεί για την δράση κατά των αρκών. Και όλο αυτό είναι πολλές φορές τμήμα ευρύτερων προγραμμάτων σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε επίσης αποφασίσει να υπάρχει ειδική κατάρτιση των συναδέλφων οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα διάφορα γεωγραφικά προγράμματα για να εξασφαλίσουμε ότι κατανοούν τα θέματα τα οποία τίθενται ιδιαίτερα για τις νάρκες. Τώρα, για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο σταθερότητος καλύτερα, από ότι κατανόησα το ερώτημά σας για τη δράση κατά των αρκών, υπάρχουν δύο κύρια τμήματα του μέσου σταθερότητος, η αντιμετώπιση των κρίσεων που καλύπτει το 70% <clears throat> της χρηματοδότησης και εδώ υπάρχουν ορισμένα προγράμματα για τη δράση κατά των αρκών, αλλά εξορισμού σχεδόν είναι μεσοπρόθεσμο με μακροπρόθεσμο πρόβλημα η αντιμετώπιση των αρκών και όχι κατεπήγον θέμα που αποτελεί κρίση. Για το τμήμα το μακροπρόθεσμο λοιπόν του μέσου σταθερότητος που είναι μονάχα το 30% του προϋπολογισμού του μέσου αυτού υπήρχε μία σιωπηρή συμφωνία όταν εγκρίθηκε αυτός ο κανονισμός ότι αυτό δεν θα αντιμετώπιζε τα θέματα της αντιμετώπισης των ναρκών και δεν θα αντικαθιστούσε την οριζόντια μεν αλλά αφοσιωμένη γραμμή του προϋπολογισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε και πάλι. Σε σχέση τώρα με το πώς θα είμαστε έτοιμοι και καλά προετοιμασμένοι για την καθαγέννη Νομίζω ότι έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στη, στα σχέδια αυτά που χρειάζονται για να έχουμε κατευθυντέ γραμμές για την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Τέλος, το ερώτημα του κ. Γκάλερ για την Αφρικανική Ένωση. Δεν έχω μπροστά μου αυτό το έγγραφο το οποίο αναφέρεται στα θέματα αυτά, αλλά νομίζω ότι στην Αφρικανική Στρατηγική, στο τομέα της ε, στρατηγικής, αναφέρεται και το θέμα της αποναρκοθέτηση και σίγουρα οι συνάδελφοί μας οι οποίοι είναι ειδικοί στα θέματα ανάπτυξης στην Αφρική γνωρίζω ότι τουλάχιστον ένας από τους πρώην συναδέλφους που κάποτε πάλι ποτέ ασχολιόταν με την οριζόντια και αφοσιωμένη γραμμή σε θέματα ανάπτυξης γνωρίζει τι ακριβώς προβλέπετε και ίσως θα μπορέσουμε μετά από αυτή τη συνάντηση να σας δώσουμε περισσότερες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανόρντεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Καλωσορίζω όλα σας τα σχόλια. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε να περάσει το μήνυμα στα κράτη-μέλη. Το πρόγραμμα συνεχίζεται διαρκεί ακόμα, δεν έχει εξαφανιστεί. Χρειάζεται και αντιμετώπιση και οικονομικούς πόρους. Εμείς τώρα με τη σειρά μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις πραγματικές ανάγκες, να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να αποφύγουμε ε, αυτή την πολιτική εκστρατεία αυτομαστίγωσης κατά τον ίδιο μας των κρατών. Θα πρέπει να εστιάσουμε στους πραγματικούς ενόχους και στην αποναρκοθέτηση και στη βοήθεια ε, στα θύματα. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί και πάλι. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα ήταν ε, η συζήτηση αυτή και το εργαστήριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μιλητές μας και τέλος θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Στις 3 η ώρα εδώ στις Βρυξέλλες σας ευχαριστώ πολύ.